Thank you. Thank you very much. Uh, Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ που ήρθατε. Αρχίζουμε τη συνεδρίαση της Σώμα ε, Επιτροπής. Έγκριση του σχεδίου ημερησία ε, διάταξη. Αν δεν έχετε παρατηρήσει, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερησία διάταξη. Ανακοινώσει δεν έχω. Να περάσουμε στο σημείο 3, ενημέρωση σχετικά με τις τρέχουσες δύο οργανικές διαπραγματεύσεις. Μπορώ να σας ενημερώσω για τις τριμερεί διαλόγους ε, πρώτο για το crowdfunding, το δεύτερο ε, στις 6 Νοεμβρίου ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο άρχισαν διαβουλεύσει για το ρόλο της ΕΣΜΑ για τις πλατφόρμες και το πεδίο εφαρμογή. Έχει γίνει πρόοδος, παραμένουν όμως όλα τα θέματα ανοιχτά προς συζήτηση. Μια τρίτη συνεδρία έχει προγραμματιστεί για τις 25 Νοεμβρίου. Έκον Envy, πλαίσιο για επενδύσεις βιώσιμες. 6 Νοεμβρίου έγινε ο δεύτερος τρίλογος οι διαπραγματεύσει. Ε, να κάνουμε την ανταλλαγή απόψεων ε, για την πρόταση ταξινόμησης και την ε, πρόταση για δημοσίευση και την εφαρμογή των δύο κανονισμών για ε, τον ορισμό του χρηματοπιστωτικού προϊόντος και του συμμετέχοντος και συμπερίληψη κοινωνικής διάστασης. Έγινε μια συζήτηση σε βάθος των άρθρων 1 ε, για το πεδίο εφαρμογής, 2 για τους ορισμούς, 3 για κριτήρια βιώσιμων και περιβαλλοντικών ε, οικονομικών δραστηριοτήτων και τέσσερα κριτήρια για ε, τις δραστηριότητες αυτές. Συμφώνησαν τα διαπραγματευόμενα μέρη να, διαπραγμα... να ε, αλλάξουν τα άρθρα 5 έως 12 σε τεχνικό επίπεδο και η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει στις 20 Νοεμβρίου. Επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 4 και 5 Νοεμβρίου. Αν δεν έχετε αντιρρήσει, παρατηρήσεις, θεωρώ ε, εγκεκριμένα τα πρακτικά των συνεδριάσεων αυτών. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 5, που είναι το βασικό θέμα μας, οικονομικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων με τον Μάριο Σεντένο, πρόεδρο της Ευρωμάδας του Eurogroup. Καλώς ορίζω τον πρόεδρο Μάριο Σεντένο. Είναι τακτικό αυτό ο διάλογο που κάναμε. Στην περασμένη κοινοβουλευτική περίοδο είχαμε ένα εξαμηνιαίο τέτοιο διάλογο. Την Άνοιξη και το φθινόπωρο κάθε φορά. Ο τελευταίο διάλογο έγινε στι 20 Νοεμβρίου 2018. Ο κύριο Σεντένο συμμετείχε επίση στην Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Εβδομάδα φέτος το Φλεβάρι. Δυστυχώς δεν είχαμε ευκαιρία να κάνουμε την άνοιξη οικονομικό διάλογο ε, λόγω ε, ε, των ευρωεκλογών και του διαλύματος που είχε προηγηθεί. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τις εργασίες στο Eurogroup και τις συστάσεις στο Συμβούλιο για την Ευρωζώνη γενικά και την υλοποίηση των συστάσεων αναχώρα για το 2019. Επίσης θα μας δώσει αυτό μια ευκαιρία να δούμε πώς βρίσκονται οι εργασίες για την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και συμπεριλαμβανομένης και της Τραπεζικής Ένωσης. Έχετε το λόγο κύριε Σεντένο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Με χαρά ε, ξανάρχομαι στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων. Ε, είναι πρώτη φορά ε, στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. και Θα ήθελα ξεκινώντας να σας συγχαρώ όλους για την εκλογή σας και εσάς κυρία Πρόεδρε για τον ε, ορισμό σας ως Πρόεδρο. Ε, και προσβλέπω σε μια αγώνιμη ανταλλαγή απόψεων και σήμερα και τους επόμενους μήνες. Σήμερα θα ήθελα πρώτα να σας μιλήσω για την οικονομική κατάσταση και το μείγμα πολιτικής και στη συνέχεια θα συνεχίσω με την ε, εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και θα κλείσω με μερικά λόγια για θεσμικά θέματα. Η Ευρωζώνη βρίσκεται ε, στο έκτο έτος και πλέον οικονομικής ανάπτυξης, αλλά η οικονομική δραστηριότητα πέρυσι έχει αρχίσει να επιβραδύνεται. Οι οικονομίες μας λειτουργούν ε, σε συνθήκες αβεβαιότητας και αντιμετωπίζουν κινδύνους που σε μεγάλο βαθμό είναι εξωτερικοί και πολιτικοί. Τι σημαίνει αυτό, ότι έχουμε ε, πετύχει να ε, συγκρατήσουμε και να επανορθώσουμε τις πηγές κινδύνου ε, την τελευταία εξαιτία εντός της Ευρωζώνης. Αλλά δεν θα πρέπει αυτό να μας κάνει να εφησυχάζουμε προσθέσαμε πάνω από 11 εκατομμύρια θέσεις εργασίας και 6 ε, συναπτά έτη οικονομικής ανάπτυξης. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις ε, μεταρρυθμίσεις ε, έτσι ώστε αυτές να είναι χωρίς αποκλεισμούς και να βελτιωθούν τα θέματα αναδιανομής υπάρχει μια βεβαιότητα και αυτή έχει ένα τίμημα ιδιαίτερα στην ε, βιομηχανία. Ε, τελευταία πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν προβλέπει ύφεση, δεν προβλέπει ύφεση ούτε σε επίπεδο μιας χώρας είτε περισσότερο. Η ε, αγορά εργασίας και παροχής υπηρεσιών έχουν δείξει ανθεκτικότητα, αλλά μπορεί να υπάρξει μετάδοση και σε αυτούς τους κλάδους. Δεν θέλω να σας θορυβήσω, αλλά ε, θα πρέπει να παρακολουθούμε τις τάσει της αγοράς και της οικονομίας. Ε, έχουμε τακτική ανταλλαγή απόψεων ε, και σχεδόν σε κάθε συνεδρίαση του Eurogroup φαίνεται ε, ε, ότι συνενούν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει να ε, συνεργάζονται όταν υπάρχει επιβράδυση και να αποφεύγουν προκυκλικές φορολογικές πολιτικές, δημοσιονομικές μάλλον. Όταν υπάρχει κάποια ύφεση δεν θα πρέπει να την επιδεινώνουμε, δεν θα πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη. Για να αποφευθεί αυτό χρειάζεται δράση εκ των προτέρων. Θα πρέπει να είναι διαφοροποιημένη στοχευμένες οι ε, δημοσιονομικές ε, ε, απαντήσεις και αντιδράσεις μας, λαμβάνοντας υπόψη το περιθώριο που έχει κάθε χώρα. Δεν θα πρέπει και πάλι να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος. Και όταν υπάρχουν ε, κίνδυνοι ε, ε, ύφηση θα πρέπει να είναι αντίστοιχη η αντίδραση. Στις συζητήσεις μας διάφορα κράτη-μέλη επίσης θεωρούν προτεραιότητα τις μεταρρυθμίσει και τις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη καθώς και στο κλίμα. Για να φτάσουμε σε αυτούς τους στόχους θα πρέπει να δημιουργήσουμε το απαραίτητο θεσμικό περιβάλλον θα ήθελα λοιπόν να έρθω στη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης που είναι ένα πρόγραμμα μακράς πνοής. Έχουμε εργαστεί εντατικά επί μια διετία τώρα. Θα αρχίσω από το δημοσιονομικό ε, μέσο για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση, BIC με δίωση, έτσι το αποκαλούμε. Ε, γνωρίζετε ότι είναι το πιο καινοτόμο στοιχείο της ΟΝΕ. Τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο συμφωνήσαμε τα βασικά ε, χαρακτηριστικά του μέσου αυτού και τη χρηματοδότησή του. Στόχο έχει να προωθεί την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση. Αλλά θα ήταν κοντόφθαλμο ε, να το δούμε μόνο κυριολεκτικά. Το θέμα δεν είναι το τι είναι αυτό το μέσο, ούτε καν τι μπορεί να γίνει, αλλά τι μπορεί να δρομολογήσει. Θα ε, ενισχύσει το πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας μας. Υπάρχει μια κλίδα που έχουμε συμφωνήσει για την κατανομή και ευνοεί χώρες ε, που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες ανταγωνιστικότητας και σύγκλησης και σωστά κάνει. Αλλά όλα τα κράτη θα επωφεληθούν από αυτό και όλοι οι πολίτες στην Ευρωζώνη. Το BIC δεν είναι ένα μέσο σταθεροποίησης ούτε σχεδιάστηκε για να είναι τέτοιο, αλλά θα φέρει πιο κοντά τις οικονομίες μας και κατά αυτόν τον τρόπο θα διευκολύνει, ε, μάλλον θα καθησυχάσει τις ανησυχίες για την ανάγκη μόνιμων μεταφορών πιστώσεων. Θα δώσει λοιπόν έτσι σταθερότητα. Όπως είπε ο Μάριο Ντράγκη στην ε, τελευταία του ομιλία πριν από λίγες εβδομάδες, Κανένας προϋπολογισμός στην ιστορία δεν ξεκίνησε με σταθεροποίηση. Το BIC είναι διαφορετικό από άλλα μέσα στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, κυρίως γιατί έχει μεγαλύτερη ευελιξία και ειδικέ ε, πρόνοιες για τη διαχείριση. Ε, θα ε, χρηματοδοτεί ε, project που θα είναι ετήσιες προτεραιότητε τη Ευρωζώνης με ευέλικτο τρόπο ανάμεσα στα διάφορα κράτη-μέλη. Επίση θα συνεισφέρει στη σταθεροποίηση των επενδύσεων επιτρέποντας χώρες να μειώσουν το ποσοστό χρηματοδοτηση σε περίοδο κρίσης. Στην αρχή η συμμετοχή θα είναι μικρή ε, των κρατών μελών. Η Φιλανδική Προεδρία ε, έχει αρχίσει την νομοθετική δουλειά σε δύο κανονισμού. Υπάρχει ευρεία στήριξη μεταξύ των κρατών, υπάρχει ειδική νομική βάση για τον ΠΙΚ, ξεχωριστή από το πρόγραμμα υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων. Ελπίζω πω οι διαπραγματεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θα ολοκληρωθούν σύντομα έτσι ώστε το εργαλείο, το μέσο δηλαδή αυτό, να αρχίσει να λειτουργεί από το 2021 και ε, υπολογίζω, στην, ε, αναμένω να μας υποστηρίξετε. Φυσικά το τελικό αποτέλεσμα θα είναι προϊόν συμβιβασμού, αλλά ο συμβιβασμός αποτελεί αναπόσταση το τμήμα τη Δημοκρατία και εδώ βρισκόμαστε στον οίκο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Τέλο, είμαι πεπισμένο ότι η θέσπιση αυτού του BIC θα μα δώσει έναν λόγο για να σκεφτούμε καλύτερα πώ να διαρθρώνουμε και πώ να προγραμματίζουμε τι ε, άτυπε ανταλλαγέ απόψεών μα. Ε, και φυσικά είμαι ανοιχτό για να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και στο μέλλον. Τώρα θα σας πω ε, και δύο λόγια σε ό,τι αφορά άλλου τομείς στους οποίους έχουμε επιτύχει πρόοδο και έχουμε επιτύχει περισσότερη ανθεκτικότητα για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Το Europro κατέληξε τον Ιούνιο σε μια συμφωνία επί τη αρχή για μια αναθεώρηση και αυτό θα επιτρέψει δηλαδή μια καλύτερη, μια πιο αποτελεσματική αξιοποίησή τη. Συγκεκριμένα δηλαδή θα υπάρχουν περισσότερα προσβάσιμα ε, προληπτικά εργαλεία ενώ θα ενισχύσουμε και το πλαίσιο της αντιμετώπισης κρίσεων. Ταυτόχρονα ε, το σύμφωνο θα ε, δημιουργήσει ε, και μια κοινή βάση ό,τι αφορά το ενιαίο Ταμείο Εξυγίασης Τραπεζών που αποτελούσε και το κομμάτι αν θέλετε, που έλειπε από την Τραπεζική Ένωση. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της οριστικοποίησης των σχετικών νομικών εγγράφων, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε με την κύρωση της, του συμφώνου του αναθεωρημένου συμφώνου για ε, σταθερότητα, πράγμα το οποίο θα πάει στο 2000, ε, στα τέλη του 2020. Σε ό,τι αφορά τώρα την Τραπεζική Ένωση, θεωρώ πω έχουμε ολοκληρώσει τι ε, απαραίτητε τεχνικέ εργασίε και τώρα βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία. Έχουμε ακολουθήσει μια σφαιρική προσέγγιση και θεωρούμε δηλαδή ότι εδώ έχουμε να κάνουμε ένα βασικό τμήμα της γενικότερης τραπεζικής ένωσης. Πέρα δηλαδή από την ασφάλιση καταθήσεων θα έχουμε και περαιτέρω ε, περγαλή όπως αυτά δηλαδή για την ενίσχυση για παράδειγμα των, της την διαφοροποίηση των κρατικών ομολόγων ε, και την μείωση της, ε, του χρηματοοικονομικού καταγερματισμού. πέρσι το Eurogroup αποφάσισε ότι θα υπάρχει μια ομάδα υψηλού επίπεδου των αναπληρωτών υπουργών οικονομικών που θα ασχολείται με αυτά τα ζητήματα και θεωρούμε πως θα επιτύχουμε πρόοδο μόνο εφόσον εξετάσουμε από κοινού όλα αυτά τα ζητήματα μέσα σε ένα συνολικό δηλαδή πακέτο, μια συνολική δέσμη ζητημάτων όπου θα υπερισχύει ενισχύσει και ένα διαλλακτικό πνεύμα. Και σε αυτό το πλαίσιο ήταν πολύ σημαντική και η πρωτοβουλία τη Γερμανία τον περασμένο μήνα που οδήγησε σε επικοδομητικέ συνομιλίε και μια διαφορετική ατμόσφαιρα, ε, μια διαφορετική διάθεση, αν θέλετε, στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα. Επίση, αναμένω να δοθεί και ένα νέο έναυσμα εδώ από τη Νέα Επιτροπή και φυσικά και από το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αρχίσουμε δηλαδή να βρισκόμαστε τώρα όλο και πιο κοντά σε ένα χάρτη πορεία σε ό,τι αφορά την έναρξη πολιτικών πλέον διαπραγματεύσεων, ώστε να υπάρξει ένα κοινό σύστημα ασφαλή καταθέσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι συνεχιζόμενε εργασίε για την εμβάθυνση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση, αυτή η δουλειά καταδεικνύει ότι τα κράτη-μέλη τη Ευρωζώνη θεωρούν ότι θα πρέπει να υπάρξει περαιτέρω ολοκλήρωση. Ε, και αυτό βέβαια είναι κάτι το οποίο μας καθησυχάζει γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση όπου η υποστήριξη απέναντι στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα την Ευρωζώνη είναι πολύ υψηλή αλλά ταυτόχρονα ο λαϊκισμός αυξάνεται και αυτός και οι διεθνείς μας ε, σχέσεις είναι ε, όλο και πιο έχουν, περιέχουν ένα και περισσότερες διαμάχες. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να διασφαλίσουμε την οικονομική ε, κυριαρχία της Ευρωζώνης ε, και την ε, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δώσουμε την πιο σημαντική απάντηση και να αντιδράσουμε στην εμπιστοσύνη των πολιτών μα μετά τι ευρωεκλογέ. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια του ε, Eurogroup τη Ευρωομάδα, έχουμε ασχοληθεί ε, ιδιαίτερα με αυτό το ζήτημα και από το 2016 αποφασίσαμε να δημοσιεύουμε τι ημερήσει διατάξει μα ε, και τα έγγραφα συνεδρίαση, τα οποία ονομάζουμε ω συνοπτικέ επιστολέ, summing up letters. θεωρώ πω αυτή η χρονική συγκυρία ήταν κατάλληλη για να κάνουμε περαιτέρω βήματα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, πάντοτε σεβόμενοι τα νομικά όρια του θεσμικού αυτού οργάνου ω ακριβώς άτυπο όργανο. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα δημοσιεύουμε τις ημερομηνίες συνεδρίασης του προπαρασκευαστικού, της προπαρασκευαστικής επιτροπής ε, του Eurogroup, του EWG και ότι επίση θα ε, ε, έχουν περισσότερες λεπτομέρειες αυτές οι συνοπτικές επιστολές και επίσης ότι θα δημιουργηθεί και ένα online, μια online σελίδα που θα περιλαμβάνει όλα αυτά τα σχετικά έγγραφα. Το τελευταίο τώρα σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ο διορισμός των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Σχετικής Τράπεζας. Γνωρίζω πως είναι ένα σημαντικό ζήτημα και γνωρίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Συμβούλιο να υπάρχει ένα short list, δηλαδή μια προκαταρκτική λίστα των υποψηφίων. Αντιλαμβάνομαι το σκεπτικό του Κοινοβουλίου, αλλά ε, γνωρίζετε πως η διαδικασία ε, επιλογής διορισμού δηλαδή έχει οριστεί στη Σύμβαση και προβλέπει δηλαδή τη συμμετοχή των θεσμικών οργάνων με συγκεκριμένη σειρά. Οπότε δεν μπορούμε εδώ να αυτοσχεδιάσουμε και δεν έχουμε και την νομική ευχαίρεια να το κάνουμε. Από τη δική μου πλευρά έχω αποφασίσει να είμαστε τελείως διαφανείς σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες που προτείνουν τα κράτη-μέλη, καθώς τις ε, δημοσιεύουμε ε, γρήγορα και άμεσα μετά ουσιαστικά από την εκνοή τη σχετική προθεσμία. Γνωρίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επίσης αναφέρει πόσο σημαντική είναι η ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων. Ε, εδώ και συμμερίζομαι την ανησυχία του Κοινοβουλίου και το τονίζω στου Υπουργού Οικονομικών κάθε φορά που προβαίνουν σε πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για υποψηφίου στο Eurogroup. Είμαι αισιόδοξο ότι τα κράτη-μέλη θα πάρουν πολύ στα σοβαρά υπόψη του το ζήτημα τη ισόρροπη εκπροσώπηση των φίλων στου μελλοντικού διορισμού και σε αυτό τον κύκλο τώρα διορισμών τη Ευρωπαϊκή Σχετική Τράπεζα βλέπουμε να κινούμαστε προ τη σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ε, πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγνωρίζει αυτή την κατεύθυνση, αυτή τη θετική εξέλιξη και θα συνεχίσει να την ενθαρρύνει ε, και στο μέλλον. Σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σεντένο. Θα ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Να υπενθυμίσω, συνηθίζουν ισχύ οι κανόνες, οι συνηθισμένοι κανόνες. Πέντε λεπτά για το κάθε μέλος. Λοιπόν, ξεκινάμε το ΕΛΚ. Ε, η Λίβια Περέιρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε του Γκρουπ, Ευρωπαίοι πολίτε ε, θεωρούν πω η Ευρωζώνη αποτελεί ένα από τα βασικά επιτεύγματα τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και γι' αυτό είναι σημαντικό ε, το να ακούμε εδώ σήμερα εδώ ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον πρόεδρο του, της Ευρωζώνης. Υπάρχει λοιπόν μια αστάθεια εδώ στη, ε, στην παγκόσμια οικονομία αλλά και βρισκόμαστε ενώπιον του Brexit. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν κάποιες φοβίες, κάποιες ανησυχίες και ενώ υπάρχουν ε, ε, πολύ συγκεκριμένε ε, προκλήσει και κατά συνέπεια είναι επίγον να δοθούν και αντίστοιχε απαντήσει. Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέο, υπάρχει ένα πρόβλημα σε ό,τι αφορά το ίδιο το χρέο, αλλά και ειδικότερα σε ό,τι αφορά και τι ε, τεράστιε διαφορέ, τι αμυσαλέ διαφορέ που υπάρχουν ανάμεσα στα διαφορετικά κράτη-μέλη. δηλαδή, ε, υπάρχουν χώρε στι οποίε τα επίπεδα είναι πολύ χαμηλότερα, ενώ σε άλλε αυτό το δημόσιο χρέο ξεπερνάει κατά 120% ε, το ΑΕΠ, όπω στην περίπτωση τη Πορτογαλία, ή 180% όπω στην Ελλάδα. Και γνωρίζετε αυτέ ποιε είναι επιπτώσει δηλαδή μια τέτοια κατάσταση. Ε, ε, οπότε θα πρέπει να αξιοποιούμε τους κάπω καλύτερε περιόδου έτσι ώστε να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι για τι περιόδου εκκρίσεων. Ιταλία Ισπανία και η Πορτογαλία, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το έλλειμμα, ξεπέρασαν το 3% κατά τελευταία χρόνια. Οπότε, ε, ενώ αυτό σημαίνει σε αυτέ τι χώρε, ενώ σε άλλε όχι, πώ θεωρείτε πω θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα τη ανισότητα διαφορετική, δηλαδή κατάσταση που ισχύει ανάμεσα στα διαφορετικά μέλη τη Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. Yes, of Okay, if you don't mind, I... Αν δεν σας πειράζει, θα απαντήσω στα πορτογαλικά. Πράγματι υπάρχουν πολύ διαφορετικές ε, καταστάσεις σε ό,τι αφορά την ιστορική εξέλιξη των δημοσίων οικονομικών των διαφορετικών κρατών μελών της Ευρωζώνης. Και αυτές οι διαφορετικές ιστορικές εξελίξεις απηχούνται φυσικά και σε ένα βασικό δίκτυο που είναι και το δημοσιοχρέο. Και γι' αυτό οι συνθήκες και τα σύμφωνα στα οποία έχουμε καταλήξει αναφέρονται και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι στις περιπτώσεις εκείνες δηλαδή όπου τα κράτη-μέλη μπορούν εφόσον ακριβώς έχουν καταφέρει να επιτύχουν συγκεκριμένους ακριβώς μεσοπρόθεσμους στόχους να ε, μην περιλαμβάνονται πλέον σε αυτούς τους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς που ενεργοποιούνται ε, στις περιπτώσεις εκείνες. Άρα λοιπόν αυτό το μείγμα των ε, δημοσιονομικών ε, πολιτικών που εφαρμόζουν έχουν ως τελικό στόχο όλα τα κράτη-μέλη μέσω πρόθεσμα να είναι σε θέση να επιτύχουν αυτούς τους στόχους σε ό,τι αφορά αυτά τα βασικά δημοσιονομικά μεγέθη. Και ακριβώς για να το επιτύχουμε χρειαζόμαστε ευελιξία αλλά και ένα από τα βασικά στοιχεία που αναφέρω εγώ, εξαιρετικά δηλαδή απαραίτητο για να φτάσουμε κάπου, η υπομονή δηλαδή, ούτως ώστε να λάβουν χώρα αυτές οι εξελίξεις που χρειάζονται το κάθε κράτος μέλος. Ε, τέτοιου είδους λοιπόν διαδικασίες είναι χρονοβόρες, ακριβώς λόγω των διαφορετικών καταστάσεων, των διαφορών που υπάρχουν ιστορικά μεταξύ των διαφορών κρατών μελών και γι' αυτό θα πρέπει να αντιμετωπίζονται και με ολοκληρωμένο τρόπο. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ακριβώς τη σημερινή χρονική συγκυρία είναι μοναδική από ιστορική άποψη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο κράτος μέλος κάτω του οποίου να έχει κινηθεί μια διαδικασία υπέρβασης ε, του ελμάτους. Και σε ό,τι αφορά αυτά τα επίπεδα ε, του χρέους, βρισκόμαστε στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε που ξεκινήσαμε δηλαδή την καταγραφή των σχετικών μεγεθών των κρατών μελών της ε, Ευρωζώνης. Νομίζω πως αυτό αποτελεί ε, και μια, ένα θετικό απολογισμό σε ό,τι αφορά τη συνολική διαδικασία δηλαδή που έχουμε ξεκινήσει. Θα πρέπει προφανώς να συνεχιστεί αυτή η δυναμική με την τήρηση των σχετικών δημοσιονομικών κανόνων, πράγμα που αποτελεί δηλαδή και υποχρέωση των ηθινόντων σε πολιτικό επίπεδο έτσι ώστε ακριβώς να διασφαλίσουμε τη συνέχιση αυτής της ιδιαίτερα θετικής εξέλιξης όπως είπα, ε, ε, και εντός και εκτός Ευρωζώνης. Και ε, πραγματικά θα πρέπει να το σημειώσουμε ότι δηλαδή ε, ενώ πριν από 2-7 χρόνια το ευρώ βρισκόταν στα πρόθυρα, αν θέλετε, τη κατάρρευση, τώρα βρισκόμαστε πολύ μακριά από εκείνο το σενάριο και θα πρέπει ακριβώ να συνεχίσουμε τη συνεργασία μα προ αυτή την κατεύθυνση. Στο Φερνάντε για του σοσιαλιστέ. Καλησπέρα σα. Καλώ ορίσατε, κύριε Σεντένο. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με τη συμφωνία του περασμένου μήνα στο Eurogroup για το μέσο αυτό, το BIC. Ε, είναι δυσδιάστατη η ερώτησή μου. Από τη μια δεν καταλαβαίνω, ακόμα δεν έχω καταλάβει την ανάγκη να μελετηθεί η υπογραφή μιας νέας διακυβερνητικής συμφωνίας. Αν ενταχθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο αυτό το μέσο, άρα οφείλει να λογοδοτεί και στο κοινοβούλιο, τότε για ποιο λόγο να υπάρχει διοργανική, μάλλον ε, διακυβερνητική συμφωνία που θα χρησιμοποιεί κονδύλια από το προϋπολογισμό για αλότριους σκοπούς και χωρίς να υπόκειται στο δημοκρατικό έλεγχο του Κοινοβουλίου δεν θα λογοδοτεί στο κοινοβούλιο, ενώ θα παίρνει χρήματα από τον προπολογισμό τον ευρωπαϊκό. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Και ένα δεύτερο πάλι που δεν μπορώ να εξηγήσω, γιατί μου φαίνεται δύσκολο. Αυτή τη στιγμή ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο συνολικό, έχει διπλό ρόλο. Και ρόλο σύγκληση μέσω των ταμείων συνοχή, των διαρθωτικών ταμείων, αλλά ταυτόχρονα βοηθάει και για την ε, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας από τον ορίζοντα 2020 και άλλα προγράμματα. Οπότε δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο τώρα υπάρχει ανάγκη να έχουμε άλλο εργαλείο στα πλαίσια του PDP, άρα περιορισμένο, για να υλοποιούμε τις ναι, ίδιες πολιτικές που έτσι και αλλιώς κάνει ήδη ο προϋπολογισμός της Ένωσης στο σύνολό του. Βελτίωση δηλαδή της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλησης. Εγώ δεν νομίζω ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται να αφαιρεί πόρους από το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πηγαίνουν μόνο στις χώρες της Ευρωζώνης τα λεφτά αυτά, χωρίς να υπάρχει ένας σταθεροποιητικός παράγων και μια λειτουργία που αυτό χρειάζεται ουσιαστικά η Ευρωζώνη. Εγώ θα ήθελα να έχει περισσότερο σταθεροποιητικό ρόλο. Γιατί για την σύγκληση και την ανταγωνιστικότητα έχουμε ήδη τον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Τι το θέλουμε το νέο μέσο. Ευχαριστώ πολύ. Thank Thank you, uh, Mr. Σας ευχαριστώ κύριε Φερνάντες για την ερώτησή σας. Η δυνατότητα ύπαρξης διακυβερνητικής συμφωνίας υπάρχει για να αποφασίσουμε για το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού. Και όχι αποφυγή ελέγχου. Δεν είναι σκοπός η αποφυγή ελέγχου από τα θεσμικά όργανα. Ελέγχου σχετικά με τη δαπάνη των χρημάτων ή πώς υλοποιούνται πολιτικές με αυτά τα χρήματα. Δύο λέξεις κλειδιά κατά την άποψή μου που είναι και οι πιο σημαντικές λέξεις και καθορίζουν την καινοτομία του BIC στη Νομισματική Ένωση, είναι διακυβέρνηση, ευελιξία. Είναι ένας νέος τρόπος διακυβέρνησης, διαχείρισης, διότι θα προσαρμόζεται στις τάσεις της Ευρωζώνης, θα προσαρμόζεται ανάγκη της Ευρωζώνης Κάτι που επεξεργαζόμαστε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Μέχρι τώρα δεν δώσαμε οικονομική διάσταση στις συστάσεις. Και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Σημαντικό για το συντονισμό πολιτικών. Πολιτικών για την Ευρωζώνη. Στόχος μας η αύξηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ από πολιτική σκοπιά είναι πολύ σημαντική διάσταση. Σημαντικότατη συνιστόσα επιτυχίας. Αναφερθήκατε στη λειτουργία της σταθεροποίησης. Έχετε πιθανότατα δίκιο. Γιατί το λέω αυτό. Μπορούμε να κινηθούμε προς μια τέτοια διάσταση αλλά είναι κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στα δημοσιονομικά μέσα που σχεδιάζουμε. Για να είμαστε άνετοι, με χρονική διάρκεια, να επαναλάβω κάτι. Κάτι που είχε πει και ο κύριος Ντράγκη. Αυτή είναι η φυσική εξέλιξη ιουδήποτε δημοσιονομικού μέσου. Το βλέπουμε αυτό ιστορικά στα δημοσιονομικά μας. Πρέπει να αισθανθούμε άνετα με αυτά που σχεδιάζουμε τώρα, να καταλάβουμε τη διάσταση αυτού που σχεδιάζουμε, τι μπορεί να καλύψει, τι μπορούμε να πετύχουμε και να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τον τομέα και μέσω των πόρων που διατίθεται και μέσω των κατάλληλων εργαλείων. Ευχαριστώ. Ο κ. Καρικάνο από το Ρινιού. Στο Πρόεδρε. Στα ισπανικά θα διαβάσω την ερώτηση, κύριε Σεντένο. Πρόεδρε Σεντένο, κοιτάξτε εδώ μια φωτογραφία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της Εκτελεστικής Επιτροπής, την περασμένη εβδομάδα. Η μόνη γυναίκα που βλέπετε εδώ στο τραπέζι είναι η κυρία Λαγκάρτ. Άλλες γυναίκες ε, βλέπουμε στα κάδρα, στους πίνακες. Πιο πολλές γυναίκες είναι στη ζωγραφική παρά στο τραπέζι. Μία είναι η γυναίκα εκεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Εμείς θέλουμε να ανανεώσουμε την Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο. Εδώ, το Renew Europe θεωρούμε ότι είναι απολύτως απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι κενό γράμμα αυτό το αίτημα ισότητας. Επειδή βάλαμε μια γυναίκα πρόεδρο και 22 άντρες από κάτω. Είναι πολλές οι γυναίκες που έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες για αυτές τις θέσεις. Δεν το αφισβητεί κανείς. Το πρόβλημα είναι διαρθρωτικό. Μας μιλήσατε για κάποιες άτυπε δράσει για να προσπαθήσετε να πείσετε τις κυβερνήσεις. Τα καταλαβαίνω αυτά που λέτε, τις άτυπε αυτές ενέργειες. Αλλά εμεί στο Renew θέλουμε περισσότερα, θέλουμε διαρθρωτικά να αλλάξει η κατάσταση, ε, διαπαντός. Και όπως γνωρίζετε, η πρότασή μας είναι να υπάρχουν δύο υποψήφοι για κάθε θέση, άνδρας και γυναίκα, για να μπορούμε πάντα να αυξάνουμε αυτή την, την ισορροπία. Οι πολίτες περιμένουν ε, ουσιαστικές δεσμεύσεις για να φτάσουμε στην ισορροπία και δεν μπορούν να ε, δεχθούν ιστοδυνικές, να δέχονται μάλλον ε, αυτή την απουσία γυναικών. Μπορούμε να υπολογίζουμε σε εσά για να φέρετε διαρθρωτικές λύσεις έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστώ κύριε Γκαρικάνο. Έχω πλήρη επίγνωση των απόψεών σας, αυτών που εξεφράστησαν και από διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου επ' αυτού. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη τις ανησυχίε σα σεβόμενοι τις αρμοδιότητες κάθε θεσμικού οργάνου και τις σχετικές, ε, σχετικούς όρους ε, περιδιορισμού προβλέπουν συνθήκες. Όπως είπα και στην αρχή, το Eurogroup αποκαλύπτει το χρονοδιάγραμμα για την επιλογή των υποψηφίων, επικρατεί διαφάνεια στη διαδικασία και είναι αρκετά αποκεντρωμένη απευθύνουμε έκκληση για υποβολή υποψηφιότητων και τα κράτη-μέλη μπορούν να παρουσιάσουν υποψηφιότητες εντός των προθεσμιών. Και ειδοποιούνται πολύ έγκαιρα τα κράτη-μέλη για τη διαδικασία. Οπότε ε, δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες αποτυχίας. Όταν καλούμε τα κράτη-μέλη να προτείνουν υποψηφίους, εγώ είχα επιμείνει από τη σημασία που έχει να επιτυγχάνεται ισορροπία των φίλων και πλουραλισμός στο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα γι' αυτό. Μπορούμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει Μπορούμε να δούμε τι γίνεται το 2019 και βλέποντας το 2019 βλέπουμε ότι έχουν γίνει κάποια σημαντικά βήματα. Όσον αφορά τις τρεις κενές θέσεις προσκάλυψη είναι έχουμε μια γυναίκα υποψήφιο που είναι θεμπρόεδρος για πρώτη φορά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για πρώτη φορά, η πιο σημαντική θέση στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και γυναίκα και άντρα υποψηφίους για τις εναπομένουσες θέσεις που είναι κενές και θα είναι κενές μέχρι το τέλος τρέχοντος έτους. Αυτό συνεπάγεται ότι ο αριθμός των γυναικών στο Συμβούλιο θα είναι ο μεγαλύτερος μέχρι τώρα στην ιστορία της ΕΚΤ. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Καλή βάση για το μέλλον και σωστή κατεύθυνση να ακολουθήσουμε. Κατανοώ τις ανησυχίες σας. Και εμένα με προβληματίζουν αυτά. Ασκήσαμε κατάλληλες πιέσεις και απέδωσαν οι πιέσεις καρπούς. Και πρέπει να συνεχίσουμε ούτω τρόπος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίγκολτ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Σεντένο, στο ίδιο θέμα και εγώ. Έχετε προσωπικά περιορισμένες δυνατότητες να κινηθείτε. Το κατανοώ. Όμως, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή την εικόνα που παρουσιάστηκε τον 21ο αιώνα. Δεν μπορούμε να βρούμε εξηγήσει εν μέρη λόγω των διορισμών εκεί που εμείς έχουμε λόγο μάλλον αφήλεται αυτή η εικόνα στο διορισμό από τι ευρωπαϊκέ κεντρικέ τράπεζε. και γι' αυτό είναι απέσια αυτή η φωτογραφία που είδαμε. Εξού και η ερώτησή μου. Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι στο Eurogroup θα ξεκινήσουν συζητήσει όσον αφορά του εθνικού διορισμού, διευθυντών κεντρικών τραπεζών. Μόνο αν έχουμε ένα δίκαιο ποσοστό γυναικών και σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να πετύχουμε ισορροπία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν μπορώ παρά να πω ότι έτσι κινδυνεύει η καλή φήμη της ΕΚΤ αν δεν αλλάξει η κατάσταση. Και το Eurogroup ε, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη. Είναι το μόνο σχήμα όπου αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα επιτυχώς. Ευχαριστώ κύριε Γκίγκολτ για την ερώτησή σας. Δεν θα σας απογοητεύσω. Επουδενή. διότι βάλετε ένα βάρος στους ώμους μου. Είναι κάτι που θα πρέπει να το εξετάσουμε από κοινού. Έτσι θα πετύχουμε αλλαγές και σε εθνικό επίπεδο, κάτι που αναφέρατε. Είναι κοινό χαρακτηριστικό του οικονομικού τομέα δυστυχώς, θα έλεγα. Η διαδικασία είναι αργοκίνητη της αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε αυτές τις καταστάσεις. Πρέπει να επιδιώξουμε βελτιώσεις, να αλλάξει όλη η ροή, να πιέσουμε προς αυτή κατεύθυνση για το μέλλον. Οι λήψεις αποφάσεων είναι αποκεντρωμένες. Οι κυβερνήσεις αποφασίζουν. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Είναι κοινή προσπάθεια. Μπορώ να σας υποσχεθώ όμως ότι το θέμα θα εξακολουθήσει να μας απασχολεί. Θα το συζητούμε όποτε υπάρχει ανάγκη τέτοιας απόφασης στο Eurogroup μαζί με τους συναδέλφους μου θα καταβάλουμε περισσότερες προσπάθειες ούτως ώστε αυτή η εικόνα να αλλάξει. Κύριος Κανονικά έχω πέντε λεπτά. Δεν διευκρινίσατε την απάντησή σας. Δεν απαντήσατε ακριβώς την ερώτησή μου. Η ερώτησή μου ποια ήταν. Μπορείτε να ξεκινήσετε συζήτηση όσον αφορά την ισορροπία των φύλων συμπεριλαμβανομένων και των διοικητών των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. Να ξεκινήσει συζήτηση όχι για τον νέο διορισμό. Είμαι σίγουρος ότι καλείται τα κράτη-μέλη να διορίσουν υποψήφιες για τις θέσεις αυτές. Το δέχομαι ότι έχετε αυτή τη δέσμευση, αλλά η ευθύνη για την εικόνα που είδαμε είναι το ζήτημα. Ερώτηση, είσαστε έτοιμος να το θέσετε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη του Eurogroup, να το συζητήσετε πώς θα αλλάξει αυτή η εικόνα, συμπεριλαμβανομένη τη ισορροπία των φύλων όσον αφορά ε, των κρατικών ε, διοικητών των κεντρικών τραπεζών. Απάντηση. Να δηλώσω ότι δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, διότι δεν έχω τα κατάλληλα μέσα στα χέρια μου στο Eurogroup να κάνω κάτι τόσο βασικό και να επηρεάσει τόσο πολύ την κάθε κυβερνητική απόφαση. Είναι ένα ζήτημα, σίγουρα. Στο επίπεδο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ θα μπορούσε να τεθεί και εκεί, εν πάση περιπτώσει. Σας διαβεβαιώ ότι Δεν θα το λησμονήσουμε το θέμα. Ούτε στην τωρινή διαδικασία, ούτε στη μελλοντική. Ούτε σε εθνικό, ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και ως ε, συντονίστης, ας το θέσω έτσι, των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, θα λάβω υπόψη μου τις ανησυχίες σας και θα τις διαβιβάσω στους Υπουργούς καταλήλως. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αντώνιο Ρινάλντι από το ID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Σεντένο, σπάνια ευκαιρία να μπορούμε να μπορείτε να μιλάτε ενώπιον ε, εκατομμυρίων ε, εκπροσώπων της, ε, των κρατών για το μέσο αυτό για τη σταθεροποίηση. Όπως είπατε και ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχε εμπλακεί ούτε διάφορα εθνικά κοινοβούλια παρά μόνο εξαιρετικά περιθωριοποιημένα. Λαμβάνονται αποφάσεις θεμελιώδους σημασία χωρίς επαρκή συζήτηση. Χρειάζεται επίσης διαφάνεια που θα δω και έτσι υπάρχει κίνδυνη αντιδημοκρατικών παρεκκλήσεων, αυταρχικών αποφάσεων και ε, δεν χρειαζόμαστε κάτι τέτοιο. Η αναδιάθρωση, η προληπτική του χρέους που γίνεται μια προϋπόθεση για την προσχώρηση σε αυτό το ταμείο ε, είναι ένα buy-in συλλογικό για εκατομμύρια πολίτες. υποχρεωτική ανάγκη για μια προληπτική προσέγγιση και, μια, και μπορεί αυτή η επέμβαση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθεροποίησης να δημιουργήσει πανικό όσον αφορά τα δημόσια αξιόγραφα και να έχει σαν ε, τελικά σαν αποτέλεσμα να έχει αυτή η πρόγνωση να αυτοπραγματοποιηθεί. Λοιπόν, μια προσπάθηση αντίδραση θα ήταν να υπάρχει χρηματοδότηση από τι αγορέ και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ευρωπαϊκό μηχανισμό σταθεροποίηση γι' αυτό. Το Ταμείο αντί να σταθεροποιεί όπω το προτείνει στην αγορά, παράδοξα θα δημιουργούσε το αντίθετο. Δηλαδή θα οδηγούσε σε αποσταθεροποίηση. Αυτή η μεταρρύθμιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού σταθεροποίηση δείχνει στου παρατηρητέ ότι γίνεται μια απόπειρα να επαναπροταθούν αυτόματοι και πιο καταναγκαστικοί μηχανισμοί ε, όταν το fiscal compact έχει αποτύχει. Από το παράθυρο προσπαθείτε να βάλετε αυτό που δεν μπήκε από την πύλη. Διότι η κυβερνητική συμφωνία όσον αφορά το fiscal compact δεν μπήκε στις συνθήκες επί των οποίων εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως προβλεπόταν εντός της πενταετίας από την ε, πρόταση αυτή. Λοιπόν, κύριε Σεντένο, έχετε αξιοποιήσει τους τεράστιους κινδύνους επαρκώς και αν ο Τζουζέπε Κόντε, πρωθυπουργό ο Ιταλό, έθεσε την όλη προβληματική ή έδωσε τη συνένεσή του χωρί να θέσει ε, καμία, κανένα βέτο. Διότι το Ιταλικό Κοινοβούλιο δεν ενημερώθηκε κατάλληλα και στι 7 του περασμένου Νοεμβρίου διάφορα μέλη του Eurogroup, των οποίων προεδρεύεται, δήλωσαν κλειστή την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού σταθεροποίηση και δεν μπορεί να υπάρχει καμία συζήτηση ή τροποποίηση πλέον. Αν η Ιταλία ή άλλη χώρα μέλος δεν μπορεί πλέον, αν τώρα δεν συμφωνεί, τι θα συμβεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γνάλντι. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθεροποίησης είναι διακυβερνητικό, διακυβερνητική συμφωνία και καλύπτεται τους κανονισμούς σύμφωνα με τη συνθήκη που δημιούργησε αυτό το μέσο του ESM. Αρκετά σημαντικό ήταν αυτό το εργαλείο για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της κρίσεως. Είναι ε, ένας προστατευτικός τείχος κατά κρίσεων που ε, αντιμετωπίσαμε εδώ και 10 χρόνια. Εάν τότε ήδη είχαμε αποφασίσει να έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο σαν το ESM, σας διαβεβαιώνω ότι θα ήμασταν πολύ επιτυχέστεροι στην αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως. Αληθεύει ότι επειδή είναι διακυβερνητική συμφωνία, εμπεριέχει συγκεκριμένους κανόνες και προβλέπει συγκεκριμένες σχέσεις με τα άλλα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Επίσης αληθεύει ότι υποβάλλονται εκθέσεις σχετικά με το ESM και τις χώρες που στο πρόγραμμα και υποβάλλονται αυτές όποτε αυτό ενδείκνυται και υποβάλλονται σχετικές εκθέσεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σας πω επίσης ότι δεν υπάρχει αυτόματη αναδιάρθρωση, καμία τέτοια αναδιάρθρωση στις ε, εφαρμοζόμενες αλλαγές στον κανονισμό περί ESM, αντιθέτως ξανασχεδιάζουμε και προτείνουμε νέους κανόνες για να αποφύγουμε επιμόλυνση διάδοση, όπως είδαμε να συμβαίνει στην κρίση 2009-2010. Είναι κάτι που απαιτεί η συζήτηση. Δεν το αμφισβητώ αυτό. Πράγματι, απαιτεί συζήτηση, ενδελεχή, τη συμμετοχή όλων σε όλα τα επίπεδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η νέα συνθήκη τον επόμενο χρόνο θα κυρωθεί από τις χώρες στο ενδεδειγμένο επίπεδο κάθε χώρας αν φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, κάτι που εύχομαι και βέβαια κατά τη διάρκεια της συζητήσεως και μετά από αυτήν αναμένουμε την ολοκλήρωση της κύρωσης σε όλα τα κράτη-μέλη και να είναι επιτυχής η διαδικασία. Πρέπει με την πάροδο κατά τη διάρκεια του επομένου έτους να παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα. Ολοκληρώνοντας την απάντησή μου, επιτρέψτε μου να σας διαβεβαιώσω λέγοντάς σας ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα θεσμικά όργανα για τη σταθερότητα. Όλοι γνωρίζουμε τις ανησυχίες σας. Να μην δημιουργηθούν αναταραχές στην αγορά για το χρέος, για το θέμα του χρέους. Και σχετικά με αυτό έχουμε μάθει από τα σφάλματα του παρελθόντος. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ο κύριος Έπινγκ από το ECR. Στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση για τη συνοχή της Ευρωζώνης. Αυτή τη στιγμή επιτάπητος έχουμε δύο θέματα. Πρώτον, το ESM, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, που είναι ένα είδος backstop, δηλαδή κάτι που μπορεί να απορροφήσει ε, ε, τους κραδασμούς όταν πτωχεύουν τράπεζες, αλλά δεν έχει τους απαραίτητους πόρους. Μετά έχουμε το EDIS που είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Ασφάλισης των Καταθέσεων που υποτίθεται ότι πρέπει να καλύπτει και τα κόκκινα δάνεια, τα μη εξυπηρετούμενα. Ποια είναι τα δύο κοινά, ότι έχουν ισχυρά χαρακτηριστικά μεταφοράς πιστώσεων και φοβούνται πολλές χώρες ε, ότι η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση θα μετατραπεί σε μία ένωση μεταφοράς χρημάτων από τη μία χώρα στην άλλη, που είναι περίπου μονόδρομος αυτό, γιατί πάντα οι ίδιοι πληρώνουν και οι ίδιοι παίρνουν. Και τώρα με τα αρνητικά επιτόκια στις χώρες που δίνουν οι ε, αποταμιευτές ή καταθέτες ε, χάνουν λεφτά και οι συνταξιούχοι υποφέρουν. Θα μπορούσατε να φανταστείτε στα πλαίσια της συνοχής της Ευρωζώνης ότι υπάρχει κοινή γνώμη σε κάποιες χώρες που δυσφορεί ή δυσανασχετεί με την κατάσταση αυτή και μπορεί να ψηφίσει ε, κόμματα που θέλουν αυτό να το σταματήσουν. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς ε, σε σχέση με τη συνοχή της Ευρωζώνης. Ευχαριστώ κύριε Έπινγκ για την ερώτησή σας αυτή. Πραγματικά είναι σημαντικές ανησυχίες τις οποίες συμμεριζόμαστε όλοι και σκεφτήκαμε όταν σχεδιάσαμε αυτά τα εργαλεία και τα μέσα και τι στόχους ε, θα πρέπει αυτά να έχουν και σε τι να αποσκοπούν. Ο γενικός στόχος αυτών των θεσμών, αυτών των μέσων και ο τρόπος με τον οποίο τα αναπτύσσουμε για να έχουμε μια τραπεζική ένωση ολοκληρωμένη είναι ακριβώς να έχουμε μια πιο σταθερή, λιγότερο κατακαιρματισμένη και σε μεγαλύτερη συνοχή ευρωζώνη. Δεν θέλω να υποτιμήσω ε, και τη διάσταση της κοινωνικής συνοχής, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι για όλες αυτές τις διαδικασίες για να, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται με τρόπο που να μην αποκλείει κανέναν και να έχει μεγαλύτερη ισορροπία στη, στην ε, αναδιανομή σε τελική ανάλυση. Αλλά επανέρχομαι στην αμεβιοποίηση και ε, στις ανησυχίες που αναφέρατε. Κοιτάξτε, νομίζω ότι κάνουμε πολύ καλή δουλειά ε, ε, για να μειώσουμε τον κίνδυνο στις οικονομίες μας. Αν κοιτάξετε και πάλι τα στοιχεία των τελευταίων ετών, θα διαπιστώσετε ότι επιτύχαμε μεγάλη μείωση των κινδύνων σε όλη την Ευρωζώνη. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της μεγαλύτερης ανθεκτικότητας που έχουμε πλέον στις οικονομίες μας μετά την ε, αθεκτικότητα ε, σε σχέση με τις ε, πιέσεις που είχαν πολλές χώρες και το σύνολο της Ευρωζώνης για τη μείωση των κινδύνων. Και αυτή η απόφαση ελήφθη ακριβώς μια στιγμή που κατανοούμε όλοι ότι ακριβώς δεν δημιουργούμε μια ένωση μεταφοράς πόρων από μια χώρα σε κάποιες χώρες σε κάποιες άλλες. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Το αντίθετο. Αυτό που θέλουμε είναι να υπάρχει εμπιστοσύνη στις διάφορες αγορές. Και να είμαστε βέβαιοι ότι όλοι οδεύουμε προς την ίδια κατεύθυνση και προχωρούμε. Στην πρώτη μου απάντηση ανέφερα όμως ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί και να μην επαναπαυόμαστε, ούτε να εφησυχάζουμε. Ακριβώς. Ε, είναι ακόμα ε, σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία πιέζουμε τα κράτη να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά ε, ε, με τρόπο ώστε να νιώθουν όλοι άνετα. Ανεφερθήκατε στα χαμηλά επιτόκια. Τα πραγματικά επιτόκια στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλά και σε πολλές χώρες εδώ και καιρό. Δεν είναι είδηση αυτό. Ισχύει εδώ και καιρό και η καλύτερη απάντηση που έχω να δώσω σε αυτή τη δυσκολία είναι η εξής. Θα πρέπει να μειώσουμε τον χρηματοπιστωτικό κατακαιρματισμό στην Ευρώπη, ε, βελτίωση των κεφαλαιαγορών ε, και επίσης οι ε, καταθέσεις μας, οι αποταμιεύσεις θα πρέπει να επενδύονται στην Ευρωζώνη σε ένα περιβάλλον ασφαλές με απόδοση. Γιατί αποδίδουν αυτές οι επενδύσεις. Και αν μπορέσουμε να προχωρήσουμε έτσι όλοι μαζί, με συνοχή, θα μειωθεί η καχυποψία, η δυσπιστία και η έλλειψη εμπιστοσύνη και θα μπορέσουμε να φτάσουμε στον τελικό μας στόχο όλων αυτών των αλλαγών, που είναι προσαρμογή στο θεσμικό μας πλαίσιο, άρα σταθερότητα γιατί αυτό είναι το ζητούμενο στην Ευρωζώνη. Ευχαριστώ. το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. 17 χρόνια της ζωής μου έχω φερώσει εδώ στο Κοινοβούλιο. Έκανα ένα διάλειμμα 5 ετών, επανήλθα και τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα πάντα έχουμε καθυστέρηση ενό τετάρτου της ώρας και πάντα η λύση δεν ενδείκνυται για τα προβλήματα που έχουμε. Ε, είμαστε σε ε, μία φάση επιβράδυνσης. Είπατε ότι μπορεί να υπάρξει και κανένα μείζον επεισόδιο. Υπάρχουν τέτοια σημεία στον ορίζοντα. Είναι γεγονός ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, έχουν περάσει τη μεγαλύτερη περίοδο ε, ανάπτυξης ε, σε όλη την ε, ιστορία τους και λέει και η γένεση στη βίβλο ότι μετά τις παχές αγελάδες έρχονται οι ισχνές. Βλέπουμε διάφορες εταιρείες να πτωχεύουν, διάφορα εργοστάσια να κλείνουν. Εδώ υπάρχουν δύο σχολές σκέψης. Ορισμένοι λέγουν ότι η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Brexit, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συμπαραμαρτούντα το πετρέλαιο, όλα αυτά τα εξωτερικά θα μας οδηγούσαν σε μια κρίση που δεν θα είναι τα κρίση ζήτησης, αλλά κρίση προσφοράς. Άλλοι πιο αισιόδοξη λέει ότι θα είμαστε σαν την Ιαπωνία. Χαμηλή ανάπτυξη, χαμηλός πληθωρισμός, χαμηλά επιτόκια. Αλλά σε χώρες όπως η δική μου Ισπανία θα έχουμε πολύ υψηλή διαρθρωτική ανεργία. Ποια είναι η δική σας απάντηση, ποια είναι τα μέτρα που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρουμε. Συμφωνώ με τον Ισπανό σοσιαλιστή συνάδελφο ότι οι διακυβερνητικοί μηχανισμοί δεν αποδίδουν. Αν θέλουμε πραγματικά να λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να πάμε στην κοινοτική μέθοδο. Στην ε, ομοσπονδιακού χαρακτήρα μέθοδο. Εναλαμβάνω, επιμένω, ποιε είναι αυτές οι λύσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται η νομισματική πολιτική δεν έχει ακόμα πολύ μπαρούτι. Έχουν τελειώσει τα πυρομαχικά. Πόσο θα μειώσουμε τα επιτόκια, ε, πώς ε, θα απαντήσουμε, με ποια μέτρα. Πώς είπε και η συνάδελφος αυτή η Πορτογαλία, Υπάρχουμε, υπάρχουν πολλές ε, χώρες εκτός από την Γερμανία, την Ολλανδία, όλοι οι άλλοι ε, είμαστε καταχρεωμένοι και έχουμε δεσμεύσεις ε, στα δημόσια οικονομικά μας. Ποιες είναι οι θεσμικές λύσεις που προτείνετε εσείς ως πρόεδρος του Eurogroup. Δεν λέω ότι θα το δεχτούν οι κυβερνήσεις, γιατί αυτά τα ξέρω. Εσείς τι θα προτείνετε. Thank you, thank you, senor Margallo, uh, for... Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαργκάλιο, για τα ερωτήματά σας. Είναι αλήθεια ότι ε, τεστάρουμε εδώ και πολύ καιρό την ανθεκτικότητα, αν θέλετε, της οικονομικής μας ανάπτυξης. Ε, δηλαδή υπάρχει πράγματι ανασφάλεια και υπάρχουν δηλαδή διαφορετικά στοιχεία τα οποία μπορούν να έχουν ε, διαφορετικές επιπτώσεις σε ό,τι αφορά την ε, εξέλιξη του παρόντος κύκλου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πάντως, η αλήθεια είναι, από το 2016 και μετά, δηλαδή από το διπομψήφισμα για το Brexit και μετά, συμπεριλαμβάνουμε όλο ένα και περισσότερο πιο πολύ αυτές τις διαστάσεις, αυτές τις δύο διαστάσεις σε ό,τι αφορά τις δικές μας δραστηριότητες, αλλά και ε, τις επιχειρήσεις δηλαδή και τη δραστηριότητά τους, αλλά και σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά, την καταναλωτική συμπεριφορά των πολιτών. Παρότι αυτά λοιπόν, ακόμα κι αν έτσι έχουν τα πράγματα, η αλήθεια είναι ότι ε, για έξι συναπτά έτη βρισκόμαστε σε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργούνται νέε θέσει ε, εργασία τη οικονομία των κρατομελών και αυτό αποτελεί απόρρια μια πιο ισορροπημένη κατάσταση σε ό,τι αφορά τη ζήτηση των οικονομιών μας αλλά και τις ε, ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις που έχουν λάβει η χώρα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωζώνης και Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την φάση της εξόδου από την οικονομική κρίση. Δεν μπορούμε να κάνουμε τα ίδια λάθη ξανά. Και γι' αυτό δεν θα πρέπει πράγματι να ε, περιμένουμε για να αντιδράσουμε σε νέα προβλήματα. Θα πρέπει να είναι προληπτική η δράση μας και νομίζω πως ε, βρισκόμαστε σε μια καλή θέση για να το κάνουμε. Γιατί σε αντίθεση ε, με κάποιες άλλες ισχυρές οικονομικές ενώσεις ανά τον κόσμο, εμείς ως ε, Ευρωζώνη έχουμε μια υγιή δημοσιονομική θέση, δηλαδή δημιουργούμε ουσιαστικά δισεκατομμύρια και τρεις εκατομμύρια ε, ευρώ ως αποταμιεύσεις ακριβώς θετικού ε, ισοζυγίου και χάρη και στις αλλαγές που έχουμε κάνει σε θεσμικό επίπεδο έχουμε ακριβώς τα καλύτερα δυνατά εργαλεία αν θέλετε στη φαρέτρα μας έτσι ώστε για να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε μια ενδεχόμενη τέτοια επιβάδυνση της οικονομίας ε, την οποία αναφέρεται. Παρότι δηλαδή δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις πηγές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αστάθεια, μπορούν να δημιουργήσουν επιβράδυνση οικονομική εδώ στην Ευρωζώνη, μπορούμε όμως να έχουμε πολιτικές οι οποίες ακριβώς δεν θα είναι προκυκλικές προς άλλους αλλά ακριβώς μια προληπτική ε, πολιτική η οποία θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια οικονομική επιβράδυνση και μείωση της ζήτησης. Κύριο ε, Περέρα τώρα για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε Μάριο Σεντένο, Πρόεδρε του Eurogroup, θα ήθελα να ξεκινήσω συγχαίροντας τις προσπάθειές σας γιατί μετά από πολλά χρόνια προσπαθειών βλέπουμε να υπάρχει μια κινητοποίηση. Κινητοποίηση δηλαδή στο επίπεδο της ε, ολοκλήρωση τη συμφωνία σε ό,τι αφορά την Τραπεζική Ένωση, αλλά και την εμβάθυνση τη Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Θα ήθελα εδώ δηλαδή να αναγνωρίσω ε, τη σημασία του νέου εργαλείου, του δημοσιονομικού δηλαδή μέσου για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση, το BIC, το οποίο μπορεί από άποψη πρικοδότηση να είναι μετριοπαθέ, αλλά παρόλα αυτά αποτελεί ένα πρώτο βήμα σε ό,τι ακριβώ ακριβώς, ε, την ε, ενίσχυση αυτών των τομέων στην Ευρωζώνη. Επίση, ε, χαιρετίζω τι προσπάθειε που γίνονται σε ό,τι αφορά πράγματι να φτάσουμε στη συμφωνία σε ό,τι αφορά ένα σύστημα ασφάλιση καταθέσεων. Βλέπουμε δηλαδή εδώ πράγματι να υπάρχει η προοπτική για να δημιουργηθεί αυτό το σύστημα, αλλά και επίση ε, με ικανοποιεί το γεγονό ότι βρισκόμαστε ακριβώς στη φάση της μεταρρύθμισης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Ε, γιατί και μέσω του ενίου Ταμείου Εξηγήσεω των Τραπεζών, με βάση αυτόν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό θα μπορέσαμε να φτάσουμε τελικά σε μια σωστή τραπεζική ένωση. Αυτά λοιπόν είναι επιτεύγματα για τα οποία σα ευχαριστώ ω πρόεδρο του Eurogroup. Αλλά παρόλα αυτά ε, δεν έχουμε ακόμα ολοκληρώσει, δεν βρισκόμαστε εκεί που θέλουμε σε ό,τι αφορά τις προσπάθειες για την σταθεροποίηση ε, της Ευρωζώνης. Ε, δηλαδή υπάρχουν κάποιες λειτουργίες τις οποίες έχουν αναλάβει τα διάφορα θεσμικά όργανα και, και η Τράπεζα, αλλά δεν έχουμε φτάσει εκεί που πρέπει ακόμα. Εκείνο λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξή. Θεωρείτε πως αυτές οι στατικές, αν θέλετε, σταθεροποίησεις εξακολουθούν να αποτελούν τμήμα της πολιτικής της Οικονομικής και Νομικής Ένωσης ε, και θα μπορούσαμε να αναμένουμε περισσότερες προσπάθειες από τη δική σας πλευρά, αν όχι στο πλαίσιο της παρούσας θητείας σας ως πρόεδρο του Eurogroup, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας δεύτερης θητείας σας. Απάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματά σας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω το εξή. Έχουμε πράγματι κάνει κάποια πρώτα σωστά, απτά και σίγουρα βήματα προς την κατεύθυνση εκείνη την οποία όλοι θεωρούμε ως σωστή. Δηλαδή την ολοκλήρωση, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση με τρόπο ε, που όλοι να νιώθουν άνετα, να νιώθουν ικανοποιημένοι με τις αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουμε κατά τη δική μου άποψη, όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε να κάνουμε ακριβώς με αυτό το σύνολο των 29 ορίμων δημοκρατιών που γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι ο ρόλος που παίζουν μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η δική μου ερμηνεία είναι ότι οι πολίτες μας ε, μετά από κάθε ευρωεκλογέ έχουν ακριβώς ενισχύσει αυτό το όραμα και αυτή την κατεύθυνση ε, την οποία υποστηρίζουμε. Και ακριβώς εμείς τώρα καλούμαστε να μεταφράσουμε, αν θέλετε, τη βούληση αυτή των πολιτών μας, όπως εκφράστηκε στις διάφορες φυγομετρήσεις και τα ευρωμαρόμετρα για το ευρώ. Να τις μεταφράσουμε λοιπόν σε συγκεκριμένα βήματα. αληθεύει το ότι για να είμαστε σε θέση να κάνουμε τα βήματα προς τη σωστή κατεύθυνση, θα πρέπει από κοινού να διασφαλίσουμε ότι θα ε, καταφέρουμε να μειώσουμε την έλλειψη εμπιστοσύνη στη δυσπιστία η οποία ε, αποτέλεσε απόρρια Τη οικονομική κρίση και η οποία συνεχίζει να παραμένει ανάμεσα στα κράτη-μέλη μας. Ε, πάντως βλέπουμε ότι πράγματι μειώνεται αυτή η δυσπιστία μέσα στους επόμενους μήνες το παρατηρούμε και χαίρομαι που και εγώ αν θέλετε προσβεύω προς τα έξω αυτήν την θετική πρόοδο για την οποία βέβαια δεν είμαι εγώ υπεύθυνο και για την οποία δεν θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει κάτι αν δεν υπήρχε ακριβώ αυτή η βούληση από την πλευρά των ε, πολιτών μα. Ε, θα συνεχίσουμε λοιπόν τι προσπάθειε που κάνουμε προ αυτή την κατεύθυνση. Ε, είναι γεγονό ότι τα δημοσιονομικά μέσα έχουν λειτουργίες οι οποίες θα πρέπει να ενσωματώσουν ακριβώς σε αυτόν τον στόχο της σταθεροποίησης. Και θεωρώ πως και στο, φουτούρο, στο, στο, μέλλον συγγνώμη, θα πρέπει να ε, συμπεριλάβουν ακόμα περισσότερο αυτή τη διάσταση της σταθεροποίησης. έτσι ώστε δηλαδή να είμαστε σε θέση να λαμβάνουμε αποφάσεις ε, για, τις, ε, για ενδεχόμενες καταστάσεις τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Ε, πάντως απαντώντας και στο ερώτημά σας, πράγματι χαιρετίζουμε και του συμβασμούς του οποίους έχουμε επιτύχει μπροστά στην κατεύθυνση. Γιατί ακριβώ αυτοί οι συμβασμοί τους οποίους επιτύχαμε αποτελούν τελικά και την απάντηση που δίνουμε εμείς ακριβώς στις επιλογές που έχουν κάνει οι πολίτες μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Λουίζα Λουίζα από το Renew. Ευχαριστώ κύριε Σεντένο. Θα ήθελα να μου πείτε περισσότερα για την ισορροπία των φύλων ή μάλλον έλλειψη ισορροπίας των φύλων. Είπατε στα αρχικά σας σχόλια ότι θα αναδείξετε το πρόβλημα αυτό της ισορροπίας των φύλων συναδέλφους και όταν σας ρώτησαν μέλη της παρούσης επιτροπής να δώσετε σαφέστερη δέσμευση. Είπατε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα έχοντας την Κριστίν Λαγκάρντ σαν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας το 2019. Για μένα το γεγονός ότι χρειαστήκαμε το 2019 για να έχουμε την πρώτη γυναίκα ε, πρόεδρο του, της ΕΚΤ, διοικητή του ΕΚΤ και είναι μόνο μια γυναίκα από 24 εκπροσώπους που κάθισαν στο τραπέζι στη φωτογραφία δείχνει ότι δεν έχουμε προχωρήσει αρκετά και έχουμε διαθωτικό πρόβλημα. Άρα απαιτείται και μια διαθωτική λύση. Σε αυτή την Επιτροπή δεν είμαστε ε, τέλειοι. Λιγότερο από 25% ε, των τακτικών μας μελών είναι γυναίκες, αλλά θέλουμε παράδειγμα, καλό παράδειγμα εκ των άνω. Και φοβούμαι ότι αυτό βαρύνει τους ε, ώμους σας και άλλους σε παρόμοιες θέσεις που έχουν επιρροή. Επίσης, να πω κάτι για την ποικιλομορφία εν γένεια. Σε αυτή την φωτογραφία λείπει. Όλοι στην εικόνα είναι λευκοί. Ξανά ρωτάω, διότι δεν ικανοποιήθηκα με τις προηγούμενες απαντήσεις σας. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Ποχήτα, για την ερώτησή σας. Κινδυνεύω να επαναλάβω αυτά που είπα, να τονίσω εκ νέου κάτι. Δεν λέω ότι θα αλλάξει η εικόνα, αυτή που δείξατε, θα αλλάξει η γενική εικόνα όμως, κατά την άποψή μου, στα θεσμικά μας όργανα, εκτός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών σε ηγετικέ θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό, πιστεύω, να συνεχίσουμε έτσι, από την πλευρά μου, και όπως βλέπω εγώ τα πράγματα θα συνεχίσω να κάνω εκστρατεία για το θέμα αυτό και θα τονίσω τις ανησυχίες που αναφέρατε μόλις τώρα. Πράγματι, το παρελθόν μας δεν μας βοηθά πολύ. Όπως είπα, το 2019 και μόνο δύο από τις τρεις τελευταίες αποφάσεις για θέσεις στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για το Συμβούλιο καλύφθηκαν από γυναίκες. Αν συνεχιστεί αυτό, θα υπάρξει δομική αλλαγή και θα αλλάξει η εικόνα που δείξατε. Υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα έχουμε καλούς υποψηφίους. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος και μετά βέβαια λαμβάνοντας υπόψη τις εκφραστήσεις ανησυχίες. Ειλικρινά, δεν βλέπω να υπάρχει άλλη λύση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την άσκηση πιέσεων όταν λαμβάνονται αποφάσεις στο μέλλον. Και έτσι αυτό που παρατηρήσαμε το 2019 να μην είναι κάτι ε, στιγμίο, αλλά κάτι που θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Χωσέ Κουσμάου από την ΚΟΕ. Thank you, Chair. I will uh, speak in Portuguese. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω πρωτοκαλικά. Κύριε Μάρα Σεντένο. Ε, ανακοινώθηκε αυτό το δημοσιονομικό μέσο με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά θα θέλαμε να γνωρίζουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εν λόγω μέσου και θα θέλαμε να γνωρίζουμε γιατί υπάρχει αυτός ενθουσιασμός για αυτό το μέσο, αν λάβουμε υπόψη μα δηλαδή τα κονδύλια αυτού του μέσου. Δηλαδή, αν εξετάσουμε εδώ το τι ακριβώς ε, συμβαίνει, ε, θα δούμε ότι το BIC θα είναι, έχει το ίμιση του δημοσιονομικού έργου σε σύγκριση με την περικοπή που έχει προβλεφθεί σε ό,τι αφορά τι πολιτικές ε, συνοχές στην Ένωση. Οπότε ένα τέτοιο ΜΠΕΚ, ένα τέτοιο μέσο δηλαδή το οποίο δεν μπορεί να ούτε καν να πλησιάσει προ το να εξισορροπήσει τι ε, περικοπές σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ ε, συνοχέ, σε τι ακριβώ τελικά θα ωφελήσει στην Ευρωζώνη. Και τώρα, εάν πράγματι βεβαιωθείτε ότι αυτά τα κονδύλια για το BIC θα αφαιρεθούν από τον ε, προπολογισμό της Ένωσης, τότε μιλάμε γιατί. Ε, αν ειδικά δηλαδή έχουν βγει από την πολιτική συνοχή, τι μιλάμε. Δεν μιλάμε καν για συμπληρωματικά κονδύλια. Μιλάμε απλά ότι έχουμε κάνει μετάθεση, αν θέλετε, ε, κονδυλίων από το ένα κομμάτι του προπολογισμού σε ένα άλλο. Χωρί να επιτυχάνουμε κάτι παραπάνω σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των συστημικών οικονομικών κρίσεων. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχουμε κανένα ε, τρόπο πραγματικό για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδου δραστηριότητε κρίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Επίση, ε, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όλε αυτέ οι προτεραιότητε τη οικονομική πολιτική δεν συνάδουν με κανέναν τρόπο με τι εκκλήσει που έχουν κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλα θεσμικά όργανα σε ό,τι αφορά την αύξηση του όγκου των επενδύσεων από την πλευρά των κρατών μελών. Γιατί αν λέμε ότι η πολιτική συνοχή που αποτελεί μια από τι βασικέ πηγέ για ακριβώ την εξαγωγή επενδύσεων, πρόκειται να περικοπτεί σε τόσο μεγάλο βαθμό, δεν είναι αυτό αποτελεσματικό μέσο για να επιτύχουμε ε, κάτι τελικά. Δηλαδή ουσιαστικά είναι αντιφατική η πολιτική που ακολουθείται εδώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Κουσμά. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο στο ευρύτερο πλαίσιο, ε, ε, μέσα, δηλαδή το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει συνδυαστεί το ε, δημοσιονομικό μέσο. Και γιατί γι' αυτό το λόγο αποτελεί ένα σημαντικό μέσο. Το δημοσιονομικό λοιπόν μέσο για την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκληση δεν αποτελεί ένα μέσο ή ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, χρηματοοικονομικό εργαλείο της πολιτικής ε, συνοχής. Δηλαδή ε, εντάσσεται σε άλλο τομέα, αλλά περιλαμβάνονται στους στόχους του ακριβώς η ενίσχυση της σύγκλησης αλλά και της ανταγωνιστικότητας των εθνικών οικονομιών. Και πώς ε, σκοπεύει να το επιχείρει αυτό με οικονομικό χαρακτήρα απαντήσεις στις προκλήσει που αναφέρονται και μέσα στο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που αφορούν τη ζώνη του ευρώ. Και είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό, δηλαδή οι συστάσεις για τη ζώνη του ευρώ έχουν ως στόχο την, το συντονισμό των πολιτικών στην Ευρωζώνη. Αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα, αλλά δεν υπήρχε ακριβώς καμία συγκεκριμένη οικονομική διάσταση, δημοσιονομική διάσταση. Αφού λοιπόν είμαστε σε θέση να δώσουμε τώρα και μια δημοσιονομική διάσταση σε αυτούς τους στόχους, αυτό καταδεικνύει ακριβώς τι σημασία που θα έχει αυτό το μέσο σε ό,τι αφορά τον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών εντό τη ζώνη του ευρώ. Ακριβώ αυτή η δυνατότητα ε, είναι που δημιουργεί το ΟΜΠΙ και αυτή τη δυνατότητα δεν θα πρέπει να την ε, χάσουμε. Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν ότι αυτό το δημοσιονομικό μέσο θα ενταχθεί στο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και βέβαια το ύψος των κοντιλίων με, το θα, με τα οποία θα προοικοδοτηθεί δεν έχει ακόμα ε, οριστικοποιηθεί. Πρόκειται δηλαδή για μια διαπραγμάτευση η οποία λαμβάνει ακόμα χώρο και θα οριστικοποιηθεί μόνο όταν θα οριστικοποιηθεί και η συνολική διαπραγμάτευση για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. και αναμένουμε ακριβώς να επιτύχει ε, περαιτέρω πρόοδο ό,τι αφορά τη δημοσιονομική διάσταση των πολιτικών μας εδώ. Τέλος, ένα σημαντικό ζήτημα και μια μοναδική πτυχή αυτού του δημοσιονομικού μέσου είναι το γεγονός ότι η διαχείρισή του γίνεται από το σύνολο των κρατών μελών της ε, ζώνης του ευρώ εστιάζοντας ακριβώς σε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Και ε, εν λόγω προτεραιότητες αυτές οι προτεραιότητες είναι ε, εκείνες οι οποίες θα οριστούν από τα ίδια τα κράτη-μέλη μέσα ε, στη, στην ζώνη του ευρώ και εκεί ακριβώς τα διάφορα κριτήρια του ζευγόνου Σταθερότητας θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Γιατί αυτό ακριβώς ε, που χρειάζεται και για την αντιμετώπιση των μελλοντικών κρίσεων είναι ακριβώς η ε, σταθεροποίηση, δηλαδή αυτή η σταθεροποιητική επιρροή που μπορεί να έχει σε επίπεδο των δημοσίων οικονομικών. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κίρτσος από το ΕΛΚΑ έχει το λόγο. Ε, έχω δύο ερωτήσεις για τον πρόεδρο κύριο Σεντένο. Η πρώτη έχει σχέση με τις ε, δηλώσεις που έκανε ο κύριος Σόλτς ε, για την εγγύηση των ευρωπαϊκών καταθέσεων. Ε, μπορείτε να μας διαφωτίσετε, είναι απλά ένα άρθρο Financial Times, είναι μια προσπάθεια, μια θέση που έχει σχέση με τα εσωκομματικά, γιατί πάνε σε συνέδριο των σοσιαλδημοκρατών, ή προφανώς θα έχετε τη σχετική πληροφόρηση. Είναι μια θέση που, έχει υιοθετήσει ή θα υιοθετήσει η γερμανική κυβέρνηση. Γιατί έχει τεράστια διαφορά ε, αν είναι το ένα ή το άλλο. Ε, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να πάμε στην εγγύηση των ε, τραπεζικών καταθέσεων, αλλά σημασία έχει ποια, είναι η άποψη της ε, γερμανικής πλευράς. Μας ενδιαφέρει πολύ. Και το δεύτερο είναι, ε, έχει σχέση με το χρέος του ελληνικό, του ελληνικού δημοσίου. Ε, το χρέος αυτό είναι τεράστιο όπως όλοι ξέρουμε, ε, αλλά στους υπολογισμούς της βιωσιμότητάς του ε, έχουν, οι υπολογισμοί αυτοί έχουν βασιστεί σε επιτόκια που τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δεν ισχύουν. Δηλαδή σε επιτόκια 4,5%, 5%, ενώ τα επιτόκια αυτή τη στιγμή που δανείζεται το ελληνικό δημόσιο, τα δεκαετή ομόλογα, είναι χαμηλότερα από το ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας που είναι γύρω στο 1,8 με 2%. Ε, ενώ με βάση τους υπολογισμούς ε, τους προηγούμενους τα επιτόκια ήταν διπλάσια ή τριπλάσια ε, από το ρυθμό ανάπτυξης. Αυτό κάνει τεράστια διαφορά σε βάθος χρόνου. Βέβαια κανείς δεν μπορεί να προφητεύσει τα επιτόκια αλλά αυτό που ξέρουμε είναι ότι οι προηγούμενοι υπολογισμοί στηρίζονται σε λάθος εκτιμήσεις θα αλλάξουν αυτοί οι υπολογισμοί. <laughs> Μας ενδιαφέρει πολύ στην Ελλάδα αυτό, γιατί έχει σχέση με το λεγόμενο ε, δημοσιονομ... πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, ουσιαστικά με τη δημοσιονομική προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κίρτσο, και για τις δύο ερωτήσεις σας. Επιτρέψτε μου να τις απαντήσω με τη σειρά. Η πρώτη ερώτηση. Βεβαίως, ακούω τα όσα λέει ο κύριος Όλαφ Σόλτς, ο συνάδελφός μου, και θεωρώ ότι είναι η θέση του Υπουργού Οικονομικών της γερμανικής κυβέρνησης. Έτσι το παρουσίασε στο Eurogroup. Άρα είναι θέση της γερμανικής κυβέρνησης. Προφανώς ε, κάνουμε διάφορες συζητήσεις και ε, στο εσωτερικό των χωρών μας και διεθνώς για αυτά τα θέματα ε, και αυτό το θέμα που αναφέρεται δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα. Χωρίς να επαναληφθώ, θα ήθελα να πω ότι ήταν πολύ σημαντική η συνεισφορά αυτή και άλλαξε ε, σε μεγάλο βαθμό το κλίμα της συζήτησης στην ε, περασμένη συνεδρίαση του Eurogroup και φυσικά προσβλέπουμε να προσθέσουμε αυτά τα στοιχεία στη συζήτηση. Αλλά πρέπει να πω ότι αυτή η συζήτηση κρατάει καιρό ήδη με διάφορες τοποθετήσεις και συνεισφορές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από την Ομάδα Εργασίας Υψηλού Επιπέδου που συστήσαμε ε, φέτος νωρίτερα και έχει ε, παρουσιάσει ήδη τρεις σημαντικές εισηγήσεις ε, για τη συζήτηση αυτή, για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου του Eurogroup. Χωρίς λοιπόν να μπω ε, σε θέματα εσωτερικής πολιτικής σκηνής στη Γερμανία και την συζήτηση, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη γερμανική κυβέρνηση για την πρόταση αυτή. Για το ελληνικό δημόσιο χρέος γνωρίζετε ότι το επιτόκιο που καταβάλει η Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερο αυτή τη στιγμή από όσα αναφέρατε. Είναι γεγονός ότι ήταν μεγάλες εξελίξεις στην αγορά ε, για την Ελλάδα και θεωρούμε ε, όλοι ότι είναι πολύ σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό και φυσικά αυτό ήταν αποτέλεσμα όλης της διαδικασίας μεταρρυθμίσεων ε, και το εκτιμούμε πάρα πολύ αυτό όλοι. Ε, αυτά είναι προσπάθειες των Ελλήνων πολιτών που καταλαβαίνουμε όλοι πόσο δύσκολο ήταν για την Ελλάδα να ε, περάσει από αυτή την προσαρμογή. Ε, κατά κάποια έννοια λοιπόν τα χαμηλά επιτόκια που βλέπετε σήμερα στις αγορές είναι κατά κάποιο τρόπο αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας που θα πρέπει να εξακολουθούμε, να την επενούμε και να τη διατηρούμε στο μέλλον. Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι λάθος εκτιμήσεις, διότι οι εκτιμήσεις έχουν να κάνουν με τον τρόπο που εκτιμάν, εκτιμούν στην αγορά τα futures, ε, τις μελλοντικέ εξελίξεις. Αλλά χρειάζεται σίγουρα ενημέρωση και επικαιροποίηση. Αναμένεται να συμβεί κάτι τέτοιο. Ε, και έχουν επιληφθεί τα θεσμικά όργανα, οι θεσμοί, και ελπίζω, και μάλλον είμαι βέβαιος, ότι ε, θα γίνει αυτό προσεχώς και επίκειται έτσι ώστε όλα αυτές τα θετικά νέα και θετικές ειδήσει να ληφθούν υπόψη. Ο Άλφρετ Σαντ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το, στην ετήσια έκθεσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο για τη μουσιονομικά το 2019 έκανε συστάσει σχετικά πώ να πλουστεύσουμε τι εξαμηνίε διαδικασίε που ακολουθούνται. Συνέστησαν την έγκριση κανόνων για δικαιολογημένε δαπάνε που συνδέεται με στόχου για τα χρέη. Λοιπόν, χρυσό Κανόνα που προστατεύει τις δημόσιες επενδύσεις, τις σχετικές δαπάνες κατά περιόδους εξηγίας οικονομικής θα πρέπει να είναι στόχοι αναχώρα που καθορίζονται και θα ενισχύεται η εφαρμογή των κανόνων με ισχυρό το διαχωρισμό μεταξύ αποφάσεων που λαμβάνονται την πολιτική και των υποκειμένων οικονομικών αξιολογήσεων. Ποια είναι η απόψή σα ε, για αυτέ τι συστάσει που έγιναν, Έχετε κάποιο πρόβλημα με κάποια συγκεκριμένη σύσταση, Μπορεί να περάσουν στο Eurogroup αυτές οι προτάσεις. Η ενίσχυση της διακυβέρνησης. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο πρότεινε ο πρόεδρος του Eurogroup θα πρέπει να έχει, απασχο... να έχει απασχόληση πλήρου χρόνου, ε, πλήρε απασχόληση να είναι τα καθήκοντά του. Ποια είναι η άποψή σα επ' αυτού. Απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Σάντ, ευχαριστώ για την ερώτησή σα. Πολύ σημαντικό θέμα. Το ανέφερα ένα-δύο φορές το θέμα σήμερα. Νομίζω ότι η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Ευθυγραμμίζεται με τις συζητήσεις που διεξήχθησαν την τελευταία διετία στο Eurogroup. Όποτε αντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα όσον αφορά εφαρμογή κανόνων μας. Να σας πω όμως ότι αντίθετα με κάποιες απόψεις που πολύ συχνά είναι αρνητικές όσον αφορά την επιτυχή εφαρμογή των παρόντων κανόνων. Αξιολογούμε τον κανόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή των λόγων κανόνων και τι αντίκτυπο έχουν οι κανόνες στη γενική προσέγγιση των δημοσιονομικών πολιτικών που ακολουθούν οι χώρες ότι όλη η αποτίμηση είναι θετική. Χρησιμοποιούμε τους κανόνες με σύνεση και ευφυΐα εφαρμόζοντας κάθε είδους ευελιξία που προβλέπεται από τους κανόνες. Κάποια φορά και πιο συχνά από το επιθυμητό, αυτοί οι κανόνες είναι πολύ δυσνόητοι και παράγουν αποτελέσματα που δεν μπορεί να τα καταλάβει και να τα προβλέψει καθαρά καθένας για κάθε χώρα. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις δυσκολίες. Γιατί αυτοί οι κανόνες το κάτω-κάτω σκοπό έχουν να διευκολύνουν τη ζωή των Υπουργών Οικονομικών μας. Και διευκολύνουν την επικοινωνία. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Να μπορεί να εξηγήσει κανείς την άμεση σχέση μεταξύ των δικών μας αποφάσεων και των ε, αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται. Υπάρχουν κάποιες απαρατήρητες μεταβλητές καμιά φορά. Δεν είναι εύκολο να εντοπιστούν. Βάση αυτής της συνεισφοράς στη συζήτηση πρέπει να πω ότι σε διάφορα επίπεδα γίνεται συζήτηση για τους κανόνες. Σύντομα, μπορούμε να συζητήσουμε ένα διαφορετικό πλαίσιο, διαφορετικό σύστημα, διαφανέστερο, πιο εύληπτο για τους κανόνες. Αυτό είναι αρκετά σημαντικό, διότι, αυτό πιστεύω εγώ, ακόμα και στην περίπτωση όπου οι κανόνες ήταν πολύ επιτυχείς όσον αφορά την προώθηση σταθερότητας των δημοσιονομικών μας, αυτό δεν γίνεται χωρίς επικρίσεις όπως βλέποντας πώς εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με μελλοντική αναθεώρηση μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση. Το συζητήσαμε σε αυτό το στάδιο, όπως σας είπα και πριν, στην αρχή, στην παρέμβασή μου. Οι επενδύσεις και επενδύσεις σε συγκεκριμένους τομείς είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη και έτσι δεν μπορούν να πλαισιώνονται μόνο εντός αυτών των κανόνων. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα βρύτερο περιθώριο. Χρειάζεται περαιτέρω συζήτηση του θέματος. Ευχαριστώ. Σβέν Γκίγκολντ από τους ε, Πράσινους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το 2019 η Ευρωζώνη έχει ακόμα ένα από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών παγκοσμίω. Και σύμφωνα με τις προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο μέλλον μπορεί να υπάρξει μείωση, αλλά αυτή θα είναι πολύ μικρή. Πιστεύετε ότι αυτό είναι βιώσιμο, καθώς αυξάνονται οι διεθνείς κραδασμοί. Θεωρείται απαραίτητο για τα κράτη-μέλη που έχουν μεγάλα πλεονάσματα να λάβουν μεγαλύτερη δράση και πώς αξιολογείται το γεγονός ότι η μεγαλύτερη χώρα σας που την χάνει να είναι η Γερμανία επέλεξε και πάλι να μην χρησιμοποιήσει το δημοσιονομικό χώρο που έχει ε, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Γκίγολτ. Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση. Ανέφερα ήδη προηγουμένως ε, τα πολύ σημαντικά πλεονάσματα ε, που έχει γενικά η Ευρωζώνη. Και νομίζω ότι είναι πραγματικά άκρο σημαντικό για μας να σχεδιάζουμε καλύτερα τους θεσμούς μας, έτσι ώστε τα πλεονάσματα αυτά να μπορούν να επανεπενδύονται στην Ευρωζώνη. Ε, και να, για να γίνει αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε έτσι περαιτέρω την Ένωση Κεφαλαιογορών και να ολοκληρώσουμε την Τραπεζική μας Ένωση. Ε, χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες θα τους ονομάσω και καμιά φορά ο πυλώνας παρά είναι ε, βαρύγδουπη λέξη γιατί υπάρχουν πολύ μικροί θεσμοί, αλλά χωρίς αυτούς τους δύο πυλώνες δεν θα μπορέσουμε ε, να προχωρήσουμε με σωστό τρόπο και να αυξήσουμε το μερίδιο του ιδιωτικού τομέα ε, στην οικονομία και στις οικονομικές και κυκλικές προσαρμογές που βλέπουμε στις οικονομίες μας. Τούτων λεχθέντων νομίζω ότι είναι σκόπιμο αυτή τη στιγμή οι χώρες ε, οι πλεονασματικές να σκεφτούν τους σωστούς τρόπους έτσι ώστε να συνεισφέρουν και εκείνες ε, στην επανεξισερώπηση της Ευρωζώνης στο σύνολό της. Υπάρχει μια διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών ε, που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το έχουμε εντοπίσει εκεί. Και πρέπει να γίνει ε, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται πώς να το πω, άλλου είδους ανισορροπίες ή εσωτερικές ε, πιέσεις σε μια χώρα αφόρητες για κάθε μία από τις χώρες αυτές που χαίρουν αυτής της κατάστασης της πλεονασματικής. Βεβαίως, έχει έρθει η ώρα να δράσουμε ε, εκ των προτέρων, όπως είπα στην ε, εισαγωγική μου τοποθέτηση, αλλά με τρόπο που να ανταποκρινόμαστε στις ανησυχίες και στις εντάσεις, ακόμα και τις κοινωνικές που μπορεί να δημιουργηθούν. Ευχαριστώ. Μια τελευταία ερώτηση. τη ΆΗ. Ο Ρόμπερτ Ρόλοντ από τους μη εγγεγραμμένους. Δύο λεπτά έχετε. Μία για την ερώτηση, μία για την απάντηση. Ευχαριστώ. Um, Ευχαριστώ ε, πολύ κύριε Σεντενό. εγώ ε, παρακολούθησα ένα ε, σεμινάριο του International Monetary Research και υπήρξαν τέσσερις κύκλοι εκεί που παρακολουθήθηκαν, δηλαδή δημόσια οικονομικά, συλλογικά δημοσιονομικά στοιχεία και δύο ακόμα στοιχεία και είδαμε ότι σε δύο από αυτά τα στοιχεία, σε ό,τι αφορά δηλαδή ειδικότερα τον επιχειρηματικό κύκλο, δεν υπήρξαν καλές εξελίξεις και και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, ένα ακόμα στοιχείο, δηλαδή ε, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει ολοένα και μεγαλύτερη απόκληση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, για παράδειγμα, ε, σε ό,τι αφορά την περίπτωση τη Γερμανία με το τεράστιο θετικό ισοζύγιο. Επίση, σε ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά. Και πάλι εδώ βλέπουμε αποκλήσει. Ε, και από εκεί και μετά, σε ό,τι αφορά τα <clears throat> συλλογικά στοιχεία, σε ό,τι αφορά ε, τα M3, τα M0 και ούτω καθεξής και πάλι εδώ δεν υπήρξε σύγκριση. Άρα λοιπόν δεν βλέπουμε σε κανένα από τα επιμέρου στοιχεία να επιτυγχάνεται αυτό ο γενικό στόχο στον οποίο αναφερθήκατε, αυτό τη σύγκληση δηλαδή. Μετά, ε, αναφερθήκατε στην αρχική σα παρουσίαση σε ε, ε μια, ένα μεγάλο πακέτο, μια μεγάλη συμφωνία σε ό,τι αφορά και την ασφάλιση των καταθέσεων. Θεωρείτε ότι αυτό οφείλεται σε μια αλλαγή τη ε, νοοτροπία τη Γερμανία ότι ε, δηλαδή αντίθετα με τι αλληλικέ ε, ε οι γερμανικέ είναι λίγο πιο ε, μετά σε ό,τι αφορά το να έχουμε τις πολιτικές τι προκυκλικές σε περίπτωση που υπάρξει μια νέα οικονομική ύφεση. Αυτό που μας λέτε ε, τι είναι, ότι αυτή δηλαδή προσπάθεια για την αποφυγή προκυκλικών πολιτικών θα πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και ποια εργαλεία θα είχατε στη διάθεσή σα Και από εκεί και μετά Εσωτερικό του, του, του ε, στόχου 2 ουσιαστικά βασίζονται σε, ε, στους ε, ε, απολογισμούς των ε, τρέχουσων, ε, συναλλαγές και στα ελλείμματα που υπάρχουν. Οπότε, πώς θα τα ερμηνεύετε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν τα πράγματα. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mr. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρόλαν. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, για να είμαι ξεκάθαρος, με τα όσα δηλαδή μας είπατε. Σε ό,τι αφορά την ε, σύγκληση που θεωρείται ότι δεν επιτεχάνεται και ότι δηλαδή αντιθέτως ε, υπάρχει απόκριση. Αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν έχουμε ε, κάποιο κάποιο αριθμό σε ό,τι αφορά το EDP. Από εκεί και μετά έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ιστορικά κρατών μελών που φτιάχνουν το MTO και επίσης έχουμε ε, ε, μεγαλύτερο, το, τον χαμηλότερο δυνατό κατακαιρματισμό ε, σε ό,τι αφορά τις ε, πολιτικέ πολιτικές μεταξύ των κρατών ε, μελών από τότε δηλαδή που ξεκίνησαν να καταγράφονται ε, τα δημοσιονομικά δεδομένα των κρατών μελών από το 1995. Σε ό,τι αφορά τώρα την ανάπτυξη Και πρώτη φορά που είναι από δύο χρόνια όλα τα κράτη-μέλη ε, είχαν ρυθμούς ανάπτυξης ανώτερους του 1,5%. Συμφωνώ όμω μαζί σα ότι δηλαδή η ανάπτυξη και οι τάσει αυτές οι ε, είναι βραδεί, οι ρυθμοί, και ότι δηλαδή δεν μπορούν ούτε να θεωρηθούν δεδομένες αυτές οι εξελίξει και ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα σε επίπεδο θεσμικών οργάνων. Και αν δούμε ε, τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, που αποτελούν ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά μια σταθερή οικονομική και νομισματική ένωση σε διαφορετικό βέβαια επίπεδο από το δικό μας. Ε, βλέπουμε ότι και εκεί η σύγκληση σε ό,τι αφορά δηλαδή αυτούς τους τομείς των δημοσίων οικονομικών είναι μια διαδικασία αργή. Και θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και τις, ε, τους ειδικούς στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Να ακολουθήσουμε αυτή την ε, περίοδο. Βέβαια υπάρχουν και κάποια τεχνικά στοιχεία σε ό,τι αφορά αυτή την ανάλυση, αλλά από εκεί και μετά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να αποφύγουμε απαντήσεις σε επίπεδο πολιτικής που είναι Και θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε την θεσμική εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, γιατί η σύγκληση δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλο τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σεντένο, ευχαριστώ και τους συναδέλφους. Νομίζω ότι εδώ ολοκληρώθηκε η συνεδρίασή μας. Υπενθυμίσω ότι η πρώτη συνεδρίαση είναι Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 18.30 και την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου μια πρωινή συνεδρίαση 9 με 12 και 30 και το απόγευμα 2.30 με 6.30. Ευχαριστώ. Γεια σας. Καλό βράδυ.